απαιτεί να λάβουμε υπόψη και τις πτυχές των τριών αυτών εκθέσεων. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ κύριε Σούλτς. Για ένα λεπτό για την ομάδα Ελευθερίας και Δημοκρατίας ο Earl of Dartmouth. Κύριε Πρόεδρε,